όπως προβλέπετε. Η Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον κανονισμό, βεβαίως, δεν ε, προβλέπεται επεξήγηση ψήφου για τα κατεπήγοντα. Από την ομάδα των φιλελευθέρων έχω λάβει ένα αίτημα να διοριστεί η κυρία Τερέσα Χιμένες Μπαρμπάτ, μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Μαγκρέτ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, καθώς επίσης και στην ε, κοινοβουλευτική διάσκεψη της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Κοινοβουλευτική συνέλευση μάλλον.